προς έγκριση την επόμενη φορά για αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις ε, τα ψηφίσματα που μόλις εγκρίναμε θα τα διαβιβάσουμε στους ε, αποδέκτες. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνει εδώ